γιατί ε, ζητείται αυτή η μείωση. Η ανησυχία μας όμως είναι η εξής. Πρώτον, συνήθως στο πλαίσιο του πολιτικού νοσομικού πλαισίου 14-20 ε, ένα τμήμα των δαπανών θα πρέπει να αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για το 2019 οι προτάσεις που γίνονται τηρούν αυτό το στόχο, αλλά όχι για τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο της περίοδου δεν θα φτάσουμε στο 20%. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας ε, έλεγξαν σε βάθος το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα μέσο όρο 20% σε όλη την περίοδο, θα πρέπει να ζητήσουμε πρόσθετες πιστώσεις 7 δισεκατομμύρια 464 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς δύσκολο, αλλά αναρωτιόμαστε, δεν θα πρέπει για την τρέχουσα ε, χρονιά, το 2018, που έχουμε ένα έλλειμμα 47,6 εκατομμυρίων ευρώ, αυτά τουλάχιστον να τα προσθέσουμε στον προπολογισμό του 2019, έτσι ώστε τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου να τηρήσουμε το συνολικό στόχο που είχε προβλεφθεί. Αυτή είναι μια ανησυχία η οποία εκφράστηκε έντονα στην ομάδα μας και σας την υποβάλλω για να την ακούστε και τη λάβετε υπόψη σας. Δεύτερη ανησυχία μας. Τα ταμεία του τίτλου του κεφαλαίου 3. Σε ό,τι αφορά την υποδοχή των προσφύγων, ε, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, τόσο πολύ έτοιμοι λειτουργικά και τόσο πολύ ε, δραστήριοι. Το βλέπετε στις διάφορες αποβιβάσεις σε Ιταλικά λιμάνια. Ε, δεν έχουμε και τόσους πολλούς όσους φανταζόμασταν. Όμως, δύο κοχαώρες ε, το Βατικανό και η Αλβανία που έδειξαν πολύ καλή διαγωγή. Και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση του Βατικανού έτσι. Μήπως θα έπρεπε όμως χώρες περιφερειακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μάλιστα κάποια στιγμή θέλουν να γίνουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα, μήπως θα έπρεπε να έχουν μια χρηματική ενίσχυση, μια οικονομική ενίσχυση, να λαμβάνουν τέτοια ενίσχυση όταν υποδέχονται πρόσφυγες. Ιδιαίτερα Προ την Αλβανία θα ήταν μια πολύ καλή χειρονομία διότι δεν είναι μέλο της Ευρωπαϊκής και αναλαμβάνει ένα τμήμα του βάρους του προσφυγικού. Μήπω λοιπόν θα έπρεπε να επιβραβευθεί οικονομικά. Σα το θέτω και αυτό υπόψη. Αυτά, Πρόεδρε. Merci. Merci pour... Euh, Πρόεδρος. Το Ταγόν. Ο κύριος Ακούσαμε ε, ήδη πολλές επικρίσεις από πλευράς των συναδέλφων. Δύσκολο, δύσκολο να διαφωνήσω μαζί τους, αδύνατο μάλλον. Δεύτερον, όπως ξέρετε είμαι λίγο ριζοσπάστης σε αυτή την επιτροπή και οποτεδήποτε κάποιος θέλει να προκαλέσει το συμβούλιο ή να του φέρει αντιρρήσεις, εγώ είμαι μπροστάρης. Μία μόνο παρατήρηση στον εισηγητή, τον οποίο θέλω και βέβαια να συγχαρώ. Ε, το έκανε και η Μόνικα Χολμάγερ και κανείς δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα από αυτήν. Αλλά θέλω να... Όχι να βάλω ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Γιατί ό,τι και να κάνει ο Ερντοάν σίγουρα δεν είναι καλές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αυτή είναι η μόνη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Κατά τα άλλα, ενωμένοι ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Merci, merci, Ευχαριστώ κύριε Τάραντ. Ε, πήραν το λόγο όλοι οι σκιοσυγητές που είναι παρόντες. Τώρα όποιο άλλος θέλει το λόγο ή όποια άλλη συνάδελφος. Ο κ. Σαρβάμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για κάτι που θα σας πω σε 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχει λόγος. Συμφωνώ με τις κριτικές που ακούστηκαν. Το Συμβούλιο δεν χρηματοδοτεί αυτά που υπόσχεται ότι θα χρηματοδοτήσει. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το σταματήσουμε. Να σας πω όμως γιατί ζήτησα το λόγο. Θέλω να σκεφτείτε το εξή. Ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για ένα ελάχιστο ποσό στο κεφάλαιο 4. Το Συμβούλιο ε, περικόπτει την διαχείριση κρίσεων. Η πολιτική προστασία και η διαχείριση κρίσεων μπορεί να λύσει πάρα πολλά τεράστια προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσπαθούν να περικόψουν, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάτι επαναστατικό προκειμένου να προληφθούν πόλεμοι και κρίσεις με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό θα πρέπει να το ανακτήσουμε. Εγώ θα προσθέτα και 5 εκατομμύρια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτό το πολύ συγκεκριμένο σημαντικό πρόβλημα. Βαλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη γενική έκθεση και τα επιμέρους. Δεν είμαι γενικός ηγετής από την ομάδα μου, όμως θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και παρατηρήσεις προς τον εισηγητή. Και σε σχέση μου σε ήδη είπε και εκείνος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κάποιες χώρες και εκτός της Ένωσης δείχνουν ελληνική και αποδέχονται τις ευρωπαϊκές αξίες. για να βοηθήσουν όχι μόνο την Ιταλία, αλλά όσε χώρε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχονται τι πιέσει ενό προβλήματο που θα έπρεπε να είναι αντικείμενο διαχείριση από κοινού. Μια τέτοια λοιπόν πρόταση μπορεί οπωσδήποτε να υποστηριχθεί, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν τις ε, ευθύνες τους, τις ηθικές τους ευθύνες, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που χάνει και ένα μεγάλο μέρος από το αρχικό πνεύμα που θα έπρεπε να διέπει το, τη δράση Θέλουμε λοιπόν εδώ να βεβαιώσω ότι θα έχουμε μεγαλύτερου αριθμού στα κονδύλια και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντο. Θέματα που όλου μα αφορούν και όπου θα πρέπει να εγκριθούν κατάλληλα κονδύλια για να μπορέσουν τα προγράμματα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως ορόσημο που θα οδηγήσουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε και κάποιες γραμμές να ενισχυθούν, κυρίως για τη Μεσόγειο, διότι θα πρέπει βεβαίω να γίνουν και διαθεσμικές διαπραγματεύσεις, όμως και το Κοινοβούλιο να έχει μια προοδευτική φωνή στα θέματα αυτά και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, γενικό προπολογισμό. Ε, βλέπουμε ότι περιλαμβάνει ένα σωρό περικοπές. Ο εισηγητής Ρούμπιχ το γνωρίζει. Διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε περικοπές με τρόπο σταθμισμένο, με τρόπο δίκαιο. Είναι τόσα τα θεσμικά όργανα που ζητούν επιπλέον περικοπές. Ας φροντίσουμε να γίνουν σωστές προσαρμογές Και σίγουρα και με τη διαδικασία του προβλεξμού του ίδιο του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, με διοικητικέ δαπάνε που θα μπορούσαν να περιοριστούν για να δώσουμε παράδειγμα σε Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι χώρε εκεί που του ζητούμε να προσαρμόσουν τον κρατικό προπολογισμό του ε, και να περιορίσουν τι δημόσιε δαπάνε, τι δαπάνε για λόγου ε, δημόσια δίκηση. Ευχαριστούμε κύριε Βάλλη. Άλλος που θα θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, συνεισηγητές για αυτή τη διεξοδική έκθεση. Περιορίζοντας τα κονδύλια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κάνουν ό,τι επιχείρησαν και στους προηγούμενους προπολογισμούς και τις σχετικές τους προτάσεις. Θα συμφωνήσω λοιπόν με όλους ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει να το επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι περικοπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες, την έρευνα, την ανάπτυξη, τον ορίζοντα 2020 και το καθεξής, τα κονδύλια αυτά μεταφέρθηκαν, μάλλον μεταφέρθηκαν ή επανακατανεμήθηκαν αλλού. Πού έχει μετατοπίσει τα κονδύλια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του θερινού διαλύματος των διακοπών έγινε πολλή κουβέντα για το Brexit. Θα πρότεινα την έκθεση αυτή να τη συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας όσο το δυνατόν συντομότερα για να έχουμε και φρέσκες πληροφορίες για το που έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις και το τι γίνεται από άποψη οικονομικών όρων. Διότι όλα αυτά θα επηρεάσουν και την ε, όλη διελκυστίντα για τον προπολογισμό το 2019 ε, και για τα επόμενα χρόνια επίσης. Ευχαριστούμε κυρία Ζουρίνη. Άλλος κανείς? Έιντερ, όχι. Όχι, οπότε προσωπικός ήθελα να πω για τα κόστη και τις περικοπές που θέλει να κάνει το Συμβούλιο το εξή. Δεν είμαι βέβαιος ότι σε αυτή τη φάση οι πολιτικές αρχές των κρατών μελών στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί ως ε, προς τις προτάσεις του Συμβουλίου οι υπάλληλοι των διαφόρων ε, ΡΕΠΕΡ εάν δεν ε, πρότειναν τις ε, συνηθισμένες περικοπές θα έπρεπε να δεχτούν επίπληξη από τους ανωτέρους τους, τους προσταμένους τους. Είναι γελίο βέβαια πολιτική διαδικασία, αλλά ήθιστε να συμβαίνει. Και πρέπει να πω ότι εάν θέλουμε να πείσουμε το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της συγκελαγής, που δεν θα είναι απλή, θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές μήνυμα εμείς ως Κοινοβούλιο και να αγωνιστούμε για κάποιες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν και μεγάλη επίκυση στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για να τι προσπιστούμε. Νομίζω τα θέματα των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών θα είναι στην καρδιά των επερχόμενων συζητήσεων. Ιδίω ε, στην φάση τη προεκλογική εκστρατεία. Έρχονται προεκλογέ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να έχουμε θέσεις που να μην είναι αμφίσιμες και να μην βασιστούν σε πρακτικές που έχουν επικρατήσει ω τώρα. Δηλαδή μηδενικό βαθμός ευρωπαϊκής ε, αλληλεγγύης και συνοχή. Αυτό φάνηκε και στις Ιταλικές εκλογέ και το αποτέλεσμά τους. Στη Σικελία το 2015 όλα αυτά με το εξελίξη εκεί ήταν απολύτως ε, δυνατόν να προβλεφθούν. Πρέπει λοιπόν η θέση μα να είναι δυνατόν να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη να μην βρούμε πολλέ προτεραιότητε να προσπιστούμε και τελικά σκοτώσουμε τι πραγματικέ προτεραιότητε. Α πούμε με την ε, Τουρκία. Μιλάμε για προένταξη. Αν κάνουμε όμω μια δημοσκόπηση στην κοινή γνώμη τη Ευρώπη για να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι και αν θέλουν την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα το κοινό μεταξύ Τουρκία ε, και του καθεστώτο ιδίω που ε, επικρατούσε και κυβερνούσε τη χώρα τη στιγμή που εγκρίθηκε η προένταξη εκεί υποστήριξη σε σχέση με το τι τώρα εκεί σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν συνέπειε όλα αυτά λοιπόν ως, προς, ως και προς τον προπολογισμό. Θα πρέπει να είμαστε ε, συνεπείς στον πολιτικό λόγο που εκφράζουμε και σε σχέση με το επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Να δούμε γιατί θα αγωνιστούμε ακριβώς, ε, γιατί το Συμβούλιο θα πρέπει να υποχρεωθεί να μας ακολουθήσει σε σχέση τουλάχιστον με αυτές τις γραμμές προτεραιότητας. και κάτι να κάνουμε ως κίνηση για τους Ευρωπαίους που υποφέρουν κάποια, ε, κάποια προσαρμογή στον προπολογισμό. Η φτώχεια επικρατεί και διωγγώνεται. Η παγκοσμιοποίηση είναι ξέφρενη και καλπάζει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βιώτη για να ολοκληρώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Με συγχωρείτε. Πρωτού δώσω το λόγο στον Γενικό Εισηγητή, ίσως να περιμένουμε και τον κύριο Μπρέζα που ε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να πω ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ δόθηκε το δικό σας γενικό εισηγητή και από τους υπόλοιπους παρεμβαίνοντας στη συζήτηση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία βασίστηκε σε αυστηρή ανάλυση των αναγκών στο υπάρχον, στο εφιστάμενο πλαίσιο και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να ε, συνδυαστούν οι διαφορετικές πολιτικές θέσεις ως προς τις προτεραιότητες και να εγκριθούν ακριβώς οι ίδιες επιθυμίες ως προς τον πολυεπολογισμό. Ως προς την Επιτροπή λοιπόν θα κοιτάξουμε να περάσουμε στις διαπραγματεύσει ε, στη φάση πριν την διαδικασία της συνδιαλλαγής δηλαδή ώστε να αποσταλεί ένα μήνυμα ε, που να δείχνει ότι η Ένωση λειτουργεί με τρόπο εύρυθμο, ότι είναι δραστήρια και ότι ως το 2019 και με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είμαστε παρόλα αυτά προετοιμασμένοι, θα έχουμε το έδαφος για την συνδιαλλαγή με αποτέλεσμα που να είναι ε, αμοιβαίως ικανοποιητικό και για τις δύο δημοσιονομικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κοιτάξει να λειτουργήσει ως παράγον διευκόλυνσης με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για τη διοικησία της συνδιαλλαγής να γίνεται σεβαστό ούτως ή άλλως και να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Ο κύριος Πρέζα λοιπόν μας είπε τα ε, τις δικές του απόψεις και τώρα ο κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις κέρυες τοποθετήσεις τους, τις κέρυες παρεμβάσεις και προτάσεις. Νομίζω ότι τις ερχόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να τα δούμε και μεταξύ μας, όχι μόνο στις επίσημες, αλλά στις άτυπες φάσεις των διαπραγματεύσεων. Καλωσορίζω όσα είπατε. Τώρα νομίζω ότι βλέπουμε καλύτερα ότι επιδιώκουμε περίπου τέτοια πράγματα όλοι. Μια-δυο συγκεκριμένες απαντήσεις όμως για ένα-δυο ζητήματα που ετέθηκαν. Και επειδή είναι περισσότερα αυτά στα οποία συμφωνούμε παρά στο που υπάρχουν διαφωνίες. Ο συνάδελφος σωστά μίλησε για την αντίθεση μεταξύ των πολιτικών των κρατών και της πολιτικής του Συμβουλίου. Εκεί ελπίζω στο Συμβούλιο να εξευρεθεί κάποιο σημείο ισορροπίας. Και συγχαίρω ήδη, ευχαριστώ μάλλον ήδη το Συμβούλιο για τις προσπάθειες συνδυασμού των πολιτικών μας προτεραιοτήτων που θα κάνει μαζί μας. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να κοιτάξουν να έχουν πολιτικέ που και τι προτεραιότητε των Ευρωπαίων πολιτών να επιδιώκουν, αλλά και τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Όλα τα θέματα που τέθηκαν είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ τον κύριο Κόλμελ, Σάβαρμα, την συνάδελφο Σούλιν για τα σχόλιά του. Να πω ότι οι επιπτώσει του Brexit δεν θα φανούν ακόμα στον προπολογισμό του 2019-2020. Είναι ένα θέμα που ευτυχώ, ευτυχώ για μένα κιόλα, δεν χρειάζεται να το επιλύσουμε τώρα με αυτή την πρόταση προπολογισμού. Θα κοιτάξουμε στι επόμενε ε, φάσει, σε μεταγενέστερα στάδια, στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο κυρίω, να βρούμε λύσει. Δύο απαντήσει στον κύριο Ντεπρέ. Πρώτο. Και εμένα αυτό με καίει που λέτε. Οι συνεργάτε σα λέτε κάνουν μια μελέτη για να δουν αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 20% επενδύσεων για το περιβάλλον. Και λέτε ότι λείπουν περίπου 7 δις. Εάν σωστά κατάλαβα, πρέπει να ζητήσουμε 7 δις παραπάνω από το Συμβούλιο. Εάν θέλετε να μου δώσετε και εμένα αυτή τη μελέτη να την κοιτάξω, εννοείται ότι μπορούμε να την θέσουμε ε, ως στόχο του Κοινοβουλίου όλου. Και ως προς την πρόταση του κ. Ντεπρέου. Εδώ δεν προσπαθώ να δώσω έμφαση σε τελικά ζητήματα. Δεν θέλω τέτοιες υποθέσεις να περάσουν στην εκθεσή μου. Όμως, εργαλεία για τις εξωευρωπαϊκές χώρες που βοηθούν την Ιταλία, την Ισπανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν τη μεταναστευτική κρίση είναι κάτι που θα μπορούσε να μα απασχολήσει. δεν μπορούμε να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μα. Όταν μιλάμε για την Αλβανία, γιατί αυτήν εννοούμε, μιλάμε για μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Μια χώρα που προσπαθεί με τεράστιε δυσκολίε να αγκιστρωθεί κάπως στην ευρωπαϊκή οικονομία και να προσχωρήσει κάποτε στην Ένωση. Έκαναν μια χειρονομία αλληλεγγύης προς την Ιταλία, διότι δέχτηκαν, μάλλον ήδη είχαν αποστείλει ε, δεκάδες χιλιάδες πολίτες τους που αποβεβάζονταν από σκάφη ε, στη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι πάντως είναι απείρως πλουσιότεροι από τους Αλβανούς για να μπορέσουν εκείνοι να λάβουν τα δικά μας βάρη τα μεταναστευτικά. Όταν μιλάμε λοιπόν για την πόλη του Βατικανού, το κράτος του Βατικανού, έκανε μια χειρονομία σημαντική, 100 πρόσφυγες στην πόλη του Βατικανού θα μείνουν στο Ιταλικό έδαφος στα πλαίσια του μεταναστευτικού συστήματος της Ιταλίας. Και πάλι ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και εύχομαι να είμαι σε θέση να είμαστε μάλλον όλοι σε θέση να έχουμε αρμονική συνεργασία και καλά αποτελέσματα στις ερχόμενες εβδομάδες. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Ευχαριστούμε που συντονίζετε την ε, όλη διαδικασία του Κοινοβουλίου ώστε να είναι αποτελεσματική. Να θυμίσω ότι οι ειδικέ επιτροπές και οι συνάδελφοι που προσωπικώς θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες πρέπει αύριο στις 12 το μεσημέρι να το κάνουν τροπολογίες ε, για τον προπολογισμό σε σχέση με την πρόταση του Συμβουλίου. 6 Σεπτεμβρίου στις 12 λίγη η προθεσμία για τις πολιτικές ομάδες. Μετά από την επενθύμηση αυτή, να πω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα γίνει την εβδομάδα 24-27 Σεπτεμβρίου. Θα ε, εργαστούμε 24, 25, 26, 27 ίσως ακόμα για τον προϋπολογισμό του 2019. Και ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε τότε και το πολιτές πλαίσιο για το 2021-2027. Και τώρα ο λόγος του συνάδελφου Χριστοφόρου για την ε, κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών και την γρήγορη και κέρια απόκριση. Κύριε Χριστοφόρου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την πολιτική μου ομάδα που με ανέθεσε να είμαι εισηγητή για το Ταμείο Αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πληρωμή προκαταβολό στο Γενικό Προπολογισμό τη Ένωση το 2019. Όπω γνωρίζετε, με πρωτοβουλία δική μα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014, αποφασίσαμε να διατίθεται ποσό ύψου 50 εκατομμυρίων ετησίω για έγκριση και άμεση αποτελεσματική καταβολή αποζημιώσεων ω προκαταβολή σε χώρε όπου υφίστανται ζημιέ ή φυσικέ καταστροφέ. Εμεί θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση ήταν πολύ εύστοχη και σημαντική, γιατί δημιουργεί τι προποθέσει να υπάρχει άμεση κινητοποίηση του Ταμείου για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των διαφόρων χωρών που υφίστανται αυτέ τι φυσικέ καταστροφέ. Ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύη δεν είναι απλά ακόμα ένα χρηματοδοτικό μέσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα μέσο που αναδεικνύει την ευαισθησία και το ανθρώπινο πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αυτό το Ταμείο οφείλουμε να το ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω. Είναι γνωστό ότι το Ταμείο έχει προπολογισμό τη τάξη των 500 εκατομμυρίων που εμεί θεωρούμε ότι σήμερα με τι συνεχιζόμενε αυξανόμενε ανάγκε ότι αυτό το ποσό πρέπει να διευρυθεί ακόμα περαιτέρω. Όμω, πρέπει να πούμε ότι αυτό το ταμείο χρειάζεται να είναι ακόμα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Και εδώ θα επισημάνω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν ανεπανόρθωτε ζημιέ και καταστροφέ. Ιδιαίτερα η Ελλάδα που είχε μέσα από τι φωνικέ πυρκαγιέ και μια τεράστια φυσική καταστροφή αλλά και εθνική τραγωδία με απώλειο ζωών. Πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι το Ταμείο θα ακούσει τη φωνή μα και άμεσα θα κινητοποιηθεί για να στηρίξει πραγματικά και γενναιόδωρα αυτήν τη χώρα που υπέστην αυτέ τι τεράστιε και πρωτόγνωρε καταστροφέ, όπω και άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υφίστανται διαρκώ εξαιτία και των κλιματικών αλλαγών αυτέ τι καταστροφέ. Μια άλλη χώρα που υπέστη και υφίσταται τα τελευταία χρόνια καταστροφή από την κλιματική αλλαγή, την ανοβρία και την λειψιδρία και θεωρείται κατάσταση έκτακτη ανάγκη είναι ολόκληρη η δική μου χώρα η Κύπρος η οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει τη μεγαλύτερη ανοβρία από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση του Ταμείου παρά τι εκκλήσει μα και πιστεύω ότι είμαστε μια ξεχωριστή περίπτωση που το Ταμείο θα μπορούσε και την Κύπρο και άλλε χώρε που υφίστανται αυτέ τι πραγματικέ χειροπιαστέ καταστροφέ από την κλιματική αλλαγή με λειψιδρία, ανοβρία, αλλά και ευρύτερη καταστροφή άμεσα το Ταμείο να ανταποκριθεί και να στηρίξει ε, την Κύπρο αλλά και άλλε χώρε που σήμερα αποτείνονται στο Ταμείο Αλληλεγγύη. Εμεί θέλουμε αυτό το Ταμείο πραγματικά να ανταποκριθεί στον την αποστολή του που δεν είναι άλλο, άμεσα, αποτελεσματικά και με ευελιξία, χωρί γραφειοκρατία, γιατί αν έχει κάτι για το οποίο κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσει, να δίνει λύσει σε μείζωνα προβλήματα σε έκτακτη ανάγκη, σε επίγουσα έκκληση των χωρών μελών για να ανταποκρίνονται στα οικονομικά και κοινωνικά του ζητήματα. Αναμένω ότι το Ταμείο άμεσα θα κινητοποιηθεί τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, αλλά πολύ περισσότερο και για τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υφίστανται διαφόρων ειδών, φυσικέ και άλλε καταστροφέ και χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Και πιστεύω ότι ω Επιτροπή οφείλουμε να πάρουμε μια απόφαση ότι μπορούμε αυτή τη δυνατότητα του Ταμείου να το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί όπω είπα, αυτό το Ταμείο αντικατοπτρίζει την κοινωνική ευαισθησία και το ανθρώπινο πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Χριστοφόρου. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις συζητητές. Κυρία Γκλουανέκ Μωρά, από τους σοσιαλιστές δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κολμέλ για το ECR. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση του. Και όντως θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδυλία. Θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ σύντομο. Θα πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κολμέλ. Οι υπόλοιποι σκιώδες εισηγητές δεν είναι εδώ παρόντες σήμερα. Άρα το λόγο θα πάρει όποιος τον επιθυμεί να εκφράσει την άποψή του τουλάχιστον. Η κυρία Κρατία Ζαμπέλ. Ε, τρία τέταρτα μπροστά από, το προβλεπόμενο χρόνο είμαστε. Ο, οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας. Ε, στηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Merci, pas δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει το λόγο. Ωραία. Κύριε Σιγητά, θέλετε ξανά το λόγο. Θέλετε ξανά το λόγο. Ε, νομίζω ότι ομόφωνα στηρίχθηκαν οι προτάσεις σας. Έχετε το λόγο. Θέλετε το λόγο. Πιστεύω ότι το μήνυμα το πολιτικό είναι πολύ ισχυρό. Όλες οι πλευρές στηρίζουν και υποστηρίζουν ότι αυτό το ταμείο να γίνει πραγματικά ταμείο αλληλεγγύης και εξορισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλεγγύης και πιστεύω ότι αυτό το ταμείο πρέπει να στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση και να είναι ακόμα πιο ενισχυμένο. Ευχαριστώ. Merci. Ainsi donc s'achève notre... εδώ η ανταλλαγή απόψεων. Οι τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, 12 ώρα το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 22-23, δεν ξέρουμε ακόμα, και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια μάλλον τη δεύτερη ε, ε σύνοδο του Δεκεμβρίου. ο λόγος στην κυρία Μάλετιτς, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, για τις κάτω χώρες και τον τραπεζικό τομέα. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι κάτω χώρες υπέβαλαν την, το αίτημά τους 23 Φεβρουαρίου 2018 μετά ε, από 1.324 απολύσεις στον τραπεζικό τομέα. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του Ταμείου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ε, η Κομισιόν ολοκλήρωσε την αξιολόγηση στις 20 Ιουλίου του 2018 και μας ε, ένα μήνα μετά, στις 20 Αυγούστου, μας έστειλε το ντοσιέ, οπότε πολύ γρήγορα το εξετάζουμε κι εμείς οι όροι του κανονισμού για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, πληρούνται. Ε, οι κάτω ζητούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, 6% δηλαδή του συνολικού κόστους που, ε, του προγραμματός τους. Πρόκειται για 20 εταιρείες του τραπεζικού τομέα και ε, οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια κρίση και την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ε, η λειτουργία των τραπεζών έχει επηρεαστεί και η κερδοφορία τους επίσης εξαιτία της ε, μείωση των επιτοκίων. οι τράπεζες χρειάστηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους, το προσωπικό τους κλείνοντας υποκαταστήματα και μετατρέποντας τις δραστηριότητε τους στο ίντερνετ. 1.324 απολύσει λοιπόν, αλλά μόνο 450 από αυτούς ε, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ε, ε επιστροφής του στην αγορά εργασίας. Οι ε, Ολλανδικές αρχές έχουν εξηγήσει ότι μόνο οι πιο ευάλωτες ομάδες θα στηριχτούν μέσω αυτών των μέτρων του Ταμείου. Αλλά οι κάτω χώρες θα καλύψουν και τους υπόλοιπους με δικά τους πόρους. Ε, στηρίζουμε αυτό το ψήφισμα ε, και την απόφαση που συνδέεται με αυτό. Ε, θα ήθελα να σας υπογραμμίσω αυτό που λέγεται στο ψήφισμα. Ε, κάνουμε έκκληση στην Κομισιόν να διασφαλίσει την πλήρη δημόσια πρόσβαση σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν καλυφθεί από το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης για λόγους διαφάνειας αλλά και προκειμένου να ανταλλάξετε καλή πρακτική και γνώση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Είναι κάτι καινούριο. Οι τράπεζες να έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Παγκοσμιοποίησης. Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Βέβαια, δεν είναι παράτυπο, αλλά θα έπρεπε ίσως να αναρωτηθούμε για το κατά πόσον θα έπρεπε να έχουν τέτοιο δικαίωμα. Το Brexit βέβαια θα μας ε, γλιτώσει από κάποιες απολύσεις στο City, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για το μέλλον. Ας προ βληματιστούμε. Χρειάζεται να, να, χρειάζεται να ε, γίνουν τουλάχιστον 500 απολύσεις για να καλυφθεί ένα κομμάτι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Άρα λοιπόν σε μια μικρή επιχείρηση δεν είναι δυνατόν. οπότε οι επιχειρήσει λένε ή θα κάνουμε πολλέ απολύσει ή καθόλου. Ε, Α προβληματιστούμε. Τροπολογίες ε, μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Ε, ψήφος στην Επιτροπή θα γίνει στις στις 24, 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου ε, και η Ολομέλεια θα εξετάσει το θέμα στην 1η Σύνοδο του Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάλετιτς. Περνάμε στο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού του 2018 είναι το υπαριθμό 5 σχέδιο αποθεματικό που σχετίζεται με τα κονδύλια που προέζονται για την Τουρκία. Ο λόγος στον Ζίκφριντ Μουρεσάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και χαίρομαι που σα ε, ξαναβλέπω και εσά και του συναδέλφου μετά το θερινό διάλειμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα προτείνει το σχέδιο ερθωτικού πρωτοπλογισμού ρυθμού 5 που περιλαμβάνει δύο στοιχεία τα οποία είναι σαφώς ε, ξεχωριστά. Το πρώτο έχει να κάνει με την Τουρκία. Όπως τα ξέρετε, όταν εγκρίναμε τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για το 2018, λάβαμε τις εξής αποφάσεις ό,τι αφορά την Τουρκία. Περικοπή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Προενταξιακού Ταμείου και βάλαμε 70 εκατομμύρια επιπλέον ε, σε αποθέματα, 70 σε εκατομμύρια για δεσμεύσει ε, για πιστώσεις και 35 για πιστώσεις πληρωμών. Γιατί καταλήξαμε ότι σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου η Τουρκία δεν κινητών προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Όταν αποφασίσαμε λοιπόν τα χρήματα αυτά να μπουν στο αποθεματικό, είπαμε ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να διατεθούν εκ νέου σε περίπτωση που υπήρχε πρόοδο σε θέματα κράτους δικαίου, ελευθερίας τύπου και το καθεξής από πλευρά της Τουρκίας. Σύμφωνα με την ετήσια έκταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκτοτε, είναι αρνητική η αιτήσια αυτή η έκθεση. Καταλήγει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι υπήρξε επαναχώρηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κράτα δικαίου, τη δημοκρατία στην Τουρκία. Άρα είναι σαφές ότι βάσει των όρων που είχαμε περιγράψει τα χρήματα του αποθεματικού δεν μπορούν να δοτηθούν εκ νέου. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν τα κονδύλια αυτά ως εξή. Τα 70 εκατομμύρια ε, πιστώσεις δεσμεύσεων. 28 εκατομμύρια προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπουν στο καταπίστευμα για την Αφρική για το, την ε, Βόρεια Αφρική για να καλυφθεί ένα κενό χρηματοδότηση που υπάρχει εκεί. 225 εκατομμύρια λείπουν το 2018 και 2019 και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις για να καλύψουμε αυτό το κενό. 42 εκατομμύρια να μπουν στο καταπιστευμένο μαντάτ για την Ιορδανία, για κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, για τους Σύριους ε, πρόσφυγες. Για τα 35 εκατομμύρια τώρα πιστώσεις πληρωμών προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάνε στην ανθρωπιστική βοήθεια για να γίνουν πληρωμές ε, λόγω της αύξησης των δεσμεύσεων στα τέλη του 2017. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά κάνει αυτές τις προτάσεις και ότι χρειάζονται τα χρήματα εκεί που, πρέπει να, που θέλει να μεταφερθούν και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των πιστώσεων δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Και γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο στοιχείο τώρα. Μία επιπλέον θέση για την ε, υπηρεσία καινοτομία. Χρειάζονται ένα ακόμα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα θέματα Wi-Fi για την Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία. Αυτή η αύξηση στο προσωπικό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον προπολογισμό της υπηρεσίας και δεν προϋποθέτει ξεχωριστές ε, πιστώσεις. Άρα για μας από δημοσιονομική άποψη είναι ουδέτερη αυτή η αύξηση προσωπικού από σπασμένο άτομο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα φύγει δηλαδή από μια παγωμένη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα ουσιαστικά θα πάει ένα άτομο στην υπηρεσία αυτή για το Wi-Fi για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν χρειάζονται επιπλέον χρήματα γιατί θα χρηματοδοτηθεί από τον προπολογισμό της υπηρεσίας. Άρα δεν έχω αντίρρηση και άρα προτείνω, κύριε Πρόεδρε, συνολικά να, προ... να... να υποστηρίξουμε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό Εισηγητή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα επιχειρήματά σα λέει ο πρόεδρο, μα οδηγούν προ την οδό τη έγκριση του σχεδίου αυτού και να δώσω το λόγο στου σκιώδει. Κύριε Καλμέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Ζίγκφριντ, τον εισηγητή, όπως πάντα. Ήταν πληρέστατος την ενημέρωσή του. Άρα δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την πρότασή σα γιατί όντω πληρούνται, μάλλον οι συνθήκε στην Τουρκία επιδεινώθηκαν δραστικά και αυτό μα οδηγεί σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Και από την άλλη, αντίστροφα, όταν υπάρχουν επιτυχή προγράμματα όπω το πρόγραμμα της δικτύωση τη σχετική υπηρεσία, προφανώ και θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε και να τα χρηματοδοτήσουμε όσο χρειάζεται για να πετύχουν ε, μεγαλύτερα αποτελέσματα. Άρα και εμείς από πλευράς μας συμφωνούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κύριο Κόλμελ. Άλλος κανείς παρακαλώ θέλει το λόγο. Νομίζω κύριε γενικά Εισηγητά ότι η έλλειψη ατόμων που να ζητούν το λόγο ε, καταδεικνύει ότι υπάρχει ομοφωνία. Ο κύριος Πρέζα. Θέλετε να μας παρουσιάσετε κάτι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να υπογραμμίσω ότι η παρουσίαση του εισηγητή και τα επιχειρήματα αν καλά το πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των κονδυλίων τα οποία είχαν προβλεφθεί το 2018 προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών και της διαχείρισης των ροών αυτών. Οπότε χαιρετίζω την πρόταση του εισηγητή να γνωμοδοτήσει θετικά και μάλιστα σε προθεσμίες που θα μας ε, επιτρέψουν να υλοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Να πω στην ότι, στην Επιτροπή μάλλον, ότι οι τροπολογίες μπορούν να καταρθούν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, στις 11 η ώρα. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσει για το θέμα αυτό την εβδομάδα 24 με 27 Σεπτεμβρίου και η Ολομέλεια θα το συζητήσει στην πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Μία ώρα νωρίς είμαστε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντοσάντος ακριβώς για το κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι η Επιτροπή Ουρομοτήπης Ουσίας με βάση επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα. 18 Οκτωβρίου θα λάβει ε, χώρα η ψηφοφορία εκεί, οπότε εμείς πρέπει να υιοθετήσουμε τη γνωμοδότησή μας στις 9 Οκτωβρίου. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων ήδη σήμερα. Ο λόγος του κύριο Ντος Σάντος. Πρόεδρε, θα ήθελα Σήμερα με τη συζήτησή μας για τον προπολογισμό το 2019 και επειδή μιλήσαμε και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κατά πάσα πιθανότητα αγγίζουμε και το θέμα που ε, καλύπτει η έκθεσή μου. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να λάβουμε κάποιες ε, αποφάσεις. Εργαστήκαμε για κατεύθυνση των διακοπών μας με τον εμπειρογνώμονά μου για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κενό ε, διάστημα. Πάντως, ε, εδώ για την ε, γνωμοδότηση, την έκθεση αυτή, καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή αυτή πιέζει ώστε το θέμα αυτό να επιληθεί γρήγορα. Σε αυτή τη φάση, τρεις ή τέσσερις παρατηρήσεις θέλω να κάνω γενικού χαρακτήρα και να αναφέρω κάποιες από τις ε, τροπολογίες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Έτσι κι τη γνωμοδότηση θα την ε, επεξεργαστούμε και τις ερχόμενες ημέρες, όμως καλό να αντιληφθούμε πολύ γρήγορα το ποιο είναι το διακύβευμα και τι μπορεί να γίνει με τους ε, προπολογισμούς, με τον προπολογισμό ως προς προσαρμογής. Η γενική αποτίμηση της πρότασης της Επιτροπής είναι θετική, διότι προσπαθεί να καθορίσει για το διάστημα μετά το 2020 το τι θα κάνει το Ταμείο αυτό και πώς θα είναι ισχυρότερο σε σχέση με τώρα. Πέραν αυτού όμως, πρόταση, στόχος της πρότασης αυτής είναι να υπάρχουν καλύτερα κριτήρια και ορισμός λύσεων που να είναι βασισμένες στη συνένεση και να είναι και αποτελεσματικές για να μπορέσουν ε, οι πολιτικές των κρατών να προσαρμοστούν αναλόγως. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει ως αποτέλεσμα των μεγάλων αφελών που αποκομίσαμε από την σκληρή δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον, των, ε, στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων Εκεί με κάποια αποτελεσματικότητα που είδαμε να πετυχάνουμε προσπαθούμε να ορίσουμε και για ένα γενικό πλαίσιο ώστε αυτός ο πυλώνας κάπως να ε, περάσει και στην πρόταση. και να καθορίσει αρχές ε, όπως η οικονομική ανάπτυξη που να είναι πιο συμμετοχική ή τις κοινωνικές πολιτικές και την πολιτική απασχόλησης σε σχέση με την θέση που θα πρέπει να ε, υιοθετήσει η Επιτροπή μας. 14 είναι αλλά ήθελα οπωσδήποτε δύο να τονίσω που μου φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση είναι μείζονος σημασίας. Πρώτον, για την ε, πρικοδότηση του Ταμείου στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταφορά χωρίς την ε, ε, ανάμεξη του Κοινοβουλίου εδώ σε κάποιες υποθέσεις. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό εφόσον δεν υπάρχουν διαφωνίες. Όμως για ειδικέ έκτακτες περιπτώσεις καλό θα ήταν να πρέπει να μπορεί να υποβάλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το, το Κοινοβούλιο. Επίσης, για το ρόλο που αναλαμβάνει εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό με τις ενισχυμένε εξουσίες που έχει στα θέματα του προπολογισμού να μπορεί τουλάχιστον υπό συγκεκριμένε ε, προποθέσει να τοποθετηθεί. Να έχει και αυτό μια κουβέντα να πει για εκταμίευση ποσών. Δεν μπορεί αυτομάτω να γίνεται πάντοτε χωρί καν να μπορεί να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην έχει δικαίωμα ψήφου και η Επιτροπή να αποφασίζει μόνη τη. Παρομοίω, κάτι που διατρέχει ολόκληρη την έκθεση και πολλέ άλλε είναι το τι θα γίνει με το βασικό προπολογισμό. Ε, για να δούμε πώ θα επηρεαστεί αναλόγω και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Θέμα είναι πώς θα ακολουθήσουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση με τις ε, διαφορές των πυλών και τις κλιματικές αλλαγές, όπως προκύπτουν και από τους σχετικούς στόχους του ΟΗΕ. Εδώ ο γενικός κανονισμός θα καθορίσει το κατά πόσον το ψήφισμά μας θα είναι ισχυρό ή όχι. Αυτές είναι οι δύο βασικές γραμμές, οι δύο βασικές τροπολογίες από τις 14 που θέλω να σχολιάσω. Θα συνεχίσουμε όμως τη δουλειά μας, ενδεχομένως να υποβληθούν κι άλλες καινούριε. Και για ένα τέτοιο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη και που ε, είναι και αρκετά απλό σε σχέση με τα υπόλοιπα που μας απασχολούν, ε, είναι ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να υποβάλουν οι ομάδες απόψεις ε, που να οδεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Για να μπορέσουμε με τους συναδέλφους, τους σκιώδεις εισηγητές, να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα και διαδικασία προπολογισμού του Ταμείου αυτού να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Το πραγματικό πρόβλημα είναι η βιάση ο επίγον χαρακτήρας ε, αυτών των ετοιμάτων. Μερικές φορές η διαδικασία διαρκεί ε, και ένα χρόνο ακόμα από τη στιγμή της κατάθεσης αίτησης. Ε, δεν μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να λαμβάνουμε γρήγορα αποφάσεις για την απελευθέρωση των κονδυλίων. Οπότε το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επιταχύνουμε Προσωπικά πιστεύω ότι το ταμείο αυτό βοηθάει πολύ τις μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν πολυάριθμες απολύσεις αλλά όχι τις πιο μικρές επιχειρήσεις. Ε, το σύστημα κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ως έναυσμα να κάνει μια επιχείρηση πολλές απολύσεις προκειμένου να ε, επωφεληθεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ε, προθεσμία για τις τροπολογίες ε, έχουν καθοριστεί 11 Σεπτεμβρίου, 18, ε, δηλαδή 6 ώρα το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε εμείς εδώ στις 9 Οκτωβρίου και η Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσει στις 18 Οκτωβρίου μάλλον. Πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Πρέζακ όμως, ποια είναι η άποψή του, πώς μπορούμε να να απλοποιήσουμε, να απλουστεύσουμε τη διαδικασία και να τις επιταχύνουμε. Κύριος Πρέζα και για την Κομισιόν. Θα ήθελα να υπογραμμίσω, να σας εκθέσω ποια είναι η προσέγγιση της Κομισιόν ως τώρα. Προκειμένου να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί στο μέτρο του δυνατού η χρήση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. όργανο αυτό είναι συμπληρωματικό για περιπτώσεις ε, που ο αριθμός των απολύσεων είναι τόσο ψηλός που χρειάζεται ευρωπαϊκή ενίσχυση. Είναι συμπληρωματικό έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται για την προσαρμογή σε διαστοτικές αλλαγές. Υπ' αυτή την έννοια η Κομισιόν έχει προτείνει ένα αριθμό βελτιώσεων. Για τις διαδικασίες προτείνουμε το εξής. Να συνδυάσουμε τις δύο υφιστάμενες παράλληλες διαδικασίες, μία για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και την διαδικασία της ε, Κινητοποίηση των κονδυλίων μέσω της διαδικασίας μεταφοράς. Προτείνουμε αυτές τις δύο να τις συνδυάσουμε σε μία πράξη, όπου η δικαιολόγηση, η αιτιολόγηση της ε, απελευθέρωσης των κονδυλίων ε, θα ε, κινητοποιεί και τις δύο διαδικασίες. Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε ποσοτικά κριτήρια κατά βάση τον αριθμό των απολύσεων που θα έχουν δικαίωμα και το ποσό το οποίο ζητείτε. Η απόφαση θα εκφράζεται σε, στο, μέσω μιας ε, συνδυασμένης πράξης και θα λαμβάνει απαραίτητο στη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα έχουν πλήρη έλεγχο της ε, απόφασης. Αλλά θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε περίπου έξι εβδομάδες κατά μέσο όρο. Επίσης, προτείνουμε να μειώσουμε το κατόφλι Εσείς προηγουμένως αναρωτηθήκατε αν οι 500 απολυμμένοι είναι ε, το πιο κατάλληλο επίπεδο. Προτείνουμε να το μειώσουμε στους 250 και πάλι βέβαια είναι σημαντικός αριθμός. Και προτείνουμε επίσης να διευρύνουμε και το πεδίο των λόγων για τους οποίους γίνονται οι απολύσεις αυτές και να συμπεριλάβουμε λόγους όπως η εισαγωγή της αυτοματοποίησης, η ψηφιοποίηση, η, με, η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές οι οποίες προτείνουμε. Ιδιαίτερα η ενοποίηση των δύο πράξεων σε μία, ε, διατηρώντας τον έλεγχο στα χέρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι η πιο σημαντική από τις αλλαγές που προτείνουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Σημειώσαμε τα όσα είπατε. Από τον Ιούλιο του 2014 βρίσκομαι σε αυτήν την Επιτροπή και κάθε φορά που κοιτάμε τέτοιου είδους εκθέσεις μπορώ να πω ότι ε, κανείς ποτέ δεν έχει κάνει κάποια πρόταση τροποποίησης της ε, ε κομισιών. Πάντοτε συμφωνούμε. Οπότε ας διερωτηθούμε. Μήπως η διαδικασία αυτή είναι υπερβολικά βαριά και θα μπορούσαν οι αποφάσεις να λαμβάνονται με πιο ελαστικό τρόπο ψυχνά, εγκρίνουμε κάτι, δίνουμε μια ενίσχυση για απολύσεις που έχουν λάβει χώρα ένα ή δύο χρόνια πριν. Αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Ντος Σάντος, θέλετε το λόγο συμπερασματικά. Πρόεδρε, ναι. Ευχαριστώ πολύ τι εσάς τον ίδιο για τα ερωτήματα και τις, προβληματισμούς που θέσατε, καθώς επίσης και την Κομισιόν. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν. Είναι βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Όμως, στην Επιτροπή μας ε, θα προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε και να την απλοποιήσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Σιγητά. Στα διάφορα, θέλει κανείς το λόγο? Όχι. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε μια μισή ώρα πριν από την προβλεπόμενη ώρα λήξης. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί και γρήγοροι. Ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Κανείς δεν ζητάει το λόγο. Κλείνουμε τη συνεδρίαση. Και τώρα θα απευθυνθώ στους συντονιστές. Η συνεδρίασή μας έχει προβλεφθεί για τις 5.30. Δηλαδή σε μία ώρα και 22 λεπτά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ήδη, αλλά μου λένε ότι ο κ. Ντεπρέ δεν θα είναι διαθέσιμος πριν τις 5. Συμφωνείτε να ξεκινήσουμε την συνάντηση των συντονιστών στις 5. Κύριος Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Στις 5. Ωραία. συντάξει συντονιστών στις 5 μετά μεσημβρία. Εδώ.